γέμισε το κοινοβούλιο κλόνου του Ταμπάιτζη και δεν αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα. Στείλτε κανένα τεχνικό σα παρακαλώ. Μάλιστα, το σημειώνουμε. Ε, και προχωρούμε στι ερωτήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πιο σύντομη σήμερα η συζήτηση αυτή, γιατί 25 λεπτά καθυστερήσαμε για λόγους διαδικαστικού. Ζητώ συγγνώμη. Θα τελειώσουμε γύρω στις 7.30 έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Μισό λεπτό, μισό λεπτό θα έχετε για τις ερωτήσεις σας σήμερα. Η πρώτη ερώτηση παριθμών 28 της κυρίας ε, Το Ο κύριος Μπαρνιά έχει το λόγο. Καλώς ορίσατε και πάλι. Παρακαλώ, απαντήστε στην ερώτηση. Ε, ευχαριστώ, Επίτροπε. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μπλινκεβιτσούτε θέτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων των συνταξιδοτικών αυτό είναι βεβαίως ε, σημαντικό θέμα για τις προκλήσεις που μας περιμένουν, καθώς και τις δυσκολίες, τα δημογραφικά προβλήματα, την κινητικότητα των εργαζομένων, την ε, κινητικότητα των πληθυσμών και γιατί τα συνταξιδοτικά ταμεία είναι και επενδυτικών ε, χαρακτηριστικών πλέον και είδαμε τι ευάλω, πόσο ευάλωτα μπορεί να είναι καθώς και η θεωρητική αντίληψη που έχουμε για τις, για πλέον. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε πρωτοβουλίε. Έχει ήδη εκφράσει κάποιου πολιτικού προσανατολισμού για το θέμα αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Και το 2010 θα παρουσιάσουμε ένα, μια πράσινη βίβλο για τις ε, συντάξεις. Ελπίζουμε ότι έτσι θα έχουμε μια πιο πλαισιωμένη συζήτηση για την ε, μεταρρύθμιση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων Επίσης, ε, την μεταρρύθμιση της οδηγίας για τις επαγγελματικέ συντάξεις και τα σχετικά επιδόματα και την αναθεώρηση της οδηγίας σε σχέση με τους κανόνες φερεγγιότητας για τα συνταξιδοτικά ταμεία. Αυτά, Πρόεδρε, ανταποκρίνονται και σε εκκλήσεις και αιτήματα του Ευρωκοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την οδηγία Solvency 2. Επίσης, ε, εδώ για θέματα που αφορούν αμέσα τους Ευρωπαίους πολίτες. Βεβαίως μας ενδιαφέρει εις όνομα της ε, επικουρικότητας να σεβαστούμε τις ε, υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Καταλαβαίνουμε ότι τα ανακατανεμητικά συστήματα είναι τα συστήματα τα οποία τα χρειάζονται ακόμα. Η κυρία Μπλίνκεβιτσούτερ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την απάντησή σας. Προσβλέπουμε στην πράσινη βίβλο που αναφέρατε. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και ανησυχεί πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, ξέρετε. Σε ορισμένα κράτη-μέλη και στη δική μου χώρα, τη Λιθουανία, οι συντάξεις μειώθηκαν πρόσφατα ε, λόγω της χρηματοοικονομικής ε, κρίσης. Ε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δίνει τόσο λίγη προσοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συντάξεις και ε, στη σταθερότητα των ε, συνταξιωτικών ταμείων και στην εγγύηση. Στη στρατηγική για το 2020 ε, λαμβάνετε τη δημογραφική κατάσταση υπόψη, την κατάσταση στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, ανησυχεί πάρα πολύ ο κόσμος. Σε 10 χρόνια θα πάρουμε συντάξεις καν. Ευχαριστώ. Επίτροπος έχει το λόγο, παρακαλώ. Euh. Κυρία μου, στο έγγραφο της στρατηγικής για το 2020, ένα έγγραφο όπου, όπου η πράσινη αύξηση, η, η συμμετοχική και πράσινη οικολογική ανάπτυξη έχει δημοσιευτεί. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε όλα τα επιμέρους ζητήματα. Έχουμε εξετάσει τα θεμελιώδη αυτά θέματα Όπω είναι και η ευθύνη μα, όπως και αυτό των συντάξεων, των συνταξιδοτικών ταμείων και τη ανεξαρτησία που πρέπει να διασφαλίσουμε για αυτά, για του Ευρωπαίου πολίτε. Ενώ ψηλών των προκλήσεων που προανέφερα. Κυρία Βλυνκεβιθούτε, σα είπα ότι τα συνταξιδοτικά ταμεία είναι σημαντικοί θεσμικοί επενδυτέ και βασίζονται στην κεφαλαιοχική συγκέντρωση των ε, κονδυλίων ε, με την ε, συμμετοχή των μελών και τις εισφορές τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα στίγμα για τα κρατημέλη και θα εργαστούμε σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας και τη βούληση πολλών θεών. Γνωρίζω πολύ καλά κάποιες τέτοιες χώρες από πολύ κοντά που θα υποστηρίξουν την παραμονή μας στην αναδιανεμητική βάση. Αυτή η δίβλος που σας προανέφερα θα δημοσιευτεί όσο το δυνατόν συντομότερα από την Επιτροπή της Προσοχής Εβδομάδας και θα έχουμε μια ευρεία συζήτηση για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Ο κύριος Όμπερ Μάιερ, παρακαλώ. Μισό λεπτό, θυμηθείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι Αυστριακός. Η Αυστρία προωθεί ε, ε, και επιδοτεί την ιδιωτική ε, συνταξιοδότηση 210 ευρώ το χρόνο. Την κεφαλαιοποίηση παρά την οικονομική κρίση θα πρέπει να προβληματιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν η συνταξιοδότηση είναι ε, καθήκον του κράτους ή όχι. Γιατί κερδοσκοπεί πολλοί κόσμος σε σχέση με αυτό. Μήπως είναι κοντόφθαλμοι ε, για να μην πω επιπόλαια η πολιτική να ε, προωθούμε και ενισχύουμε κάποιους ιδιώτες χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς να ξέρουμε τι ταμεία είναι αυτά. Γιατί όταν χρεοκοπούν αυτοί και επιτοχεύουν, έρχεται πάλι το κράτος να υποστηρίξει τη συντάξη. Ευχαριστώ. Επίτροπος. Ο πρόεδρος Μπαρόζο από αυτή τη θέση προ λίγου είχε τη δυνατότητα να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις για το ευρύ αυτό θέμα των ε, χρηματοοικονομικών ε, συναλλαγών. Εσείς αναφέρατε την κερδοσκοπία. Εγώ μπορώ να σας πω ως υπεύθυνο Ευρωπαίος Επίτροπος για τέτοια θέματα, για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες και ω προ την ε, διευθέτηση των ζητημάτων αυτών και τη ρύθμιση την ευρωπαϊκή, να σα πω ότι δεν θα αφήσουμε κανένα προϊόν, καμία, καμία επικράτεια, καμία αγορά εκτός εφιούς εποπτείας και αποτελεσματικής διευθέτησης και διακανονισμών. Όλες αυτές οι αγορές με τα διάφορα προϊόντα που συμπεριλαμβάνουν θα καλυφθούν από τις προσπάθειες που εμείς ήδη καταβάλουμε. Με το πακέτο εποπτείας που βρίσκεται υπό συζήτηση και με τις διαδοχικές αναθεωρήσεις οδηγιών, ιδίως της οδηγίας ε, για τα διάφορα παράγωγα. Θα έχουμε αυστηρούς κανόνες και κανένα από αυτά τα προϊόντα, καμία αγορά δεν θα μείνει εκτός του πλαισίου εποπτείας που θα διαμορφώσουμε, των αναγκών και απαιτήσεων διαφάνειας και εφιούς διαχείρισης. Uh, Μία επιπλέον ερώτηση. Κυρία Τσικάου, μισό λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στα γαλλικά η κυρία Τσεκάου και τώρα στα ρουμανικά. Υπάρχει στρατηγική ε, μακροπρόθεσμη σε ό,τι αφορά τα συνταξιωτικά συστήματα και τα ιδιωτικά και τα δημόσια. Τι εννοώ. Στη δεκαετία του 70 είχαμε πολύ μεγάλη γεννητικότητα και σε 30 χρόνια ε, οι άνθρωποι αυτοί θα βγουν στη σύνταξη. Σήμερα η γεννητικότητα είναι πολύ χαμηλή. Έχει καταβαραθρωθεί. Και όσοι γεννιούνται σήμερα, μετά από 30 χρόνια, θα εργάζονται μένα αλλά δηλαδή δεν θα μπορούν να διατηρούν τα ταμεία με τις εισφορές του. Και τι θα γίνει λοιπόν, έχετε την πρόθεση να λάβετε τίποτα μέτρα για την πραγματική αναθεώρηση των συστημάτων μακροπρόθεσμα υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών και με τρόπο αηφόρο και βιώσιμο. Ευχαριστώ. Euh, Κυρία Τσικάου, ήδη από την πρώτη φράση της παρέμβασής μου, Σα είπα ότι αυτό είναι μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει, πέραν δηλαδή τη κινητικότητα, μια από τι βασικέ μα προκλήσει για το μέλλον είναι το δημογραφικό θέμα. Βεβαίω όλοι μα ενδιαφέρει να έχουμε εδώ μια συζήτηση συγκρίνοντα του διάφορου όρου του προβλήματο. Ακόμη και αν δεν είναι μια από τι πρώτε ευρωπαϊκέ αρμοδιότητε το δημογραφικό ζήτημα, αλλά όλου μα αφορά και με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση. Η ήπειρο μα είναι ίσως η γυρότερη πύρος του κόσμου και χάνει συνεχώς πληθυσμό εφόσον το ποσοστό γεννήσεων δεν ανανεώνεται σε σχέση με τις ανάγκες της Υπήρου. Είναι λοιπόν ένα πλαίσιο σοβαρό, ίσως και ανησυχητικό αυτό στο οποίο πρέπει να εργαστούμε και ιδίως για το ζήτημα των συντάξεων και την ανεξαρτησία που θέλουμε να διασφαλίσουμε για, τα, για την ίδια τη σύνταξη ως έννοια, αυτή καθεαυτή. Θεωρώ λοιπόν ότι η πράσινη βίβλος είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, είναι κατάλληλη χρονική στιγμή επίση. Θα μπορέσετε να εργαστείτε για τα θέματα αυτά, να συζητήσετε, να δείτε ποιε θα είναι οι εθνικέ αρμοδιότητε για τι συντάξει, τι μπορεί να γίνει επίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίω για τα ιδιωτικά συνταξιδοτικά ταμεία και το κατά πώς αυτά διαρθρώνονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Κανένα από τα θέματα αυτά δεν θα το αφήσουμε απ' έξω από τις προτάσεις που θα περιλαμβάνει η πράσινη βίβλος όπως σας είπα, θα δημοσιευθεί εντός των ερχόμενων μηνών. Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπα. Η επόμενη ερώτηση, η παριθμόν 29 από τον Σον Κέλλη, για τα ασφαλιστικά συστήματα έναντι πλημμύρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πίτροπα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Σον Κελί κάνει μια ερώτηση που συνδέεται με μια τραγική πτυχή της επιχειρότητας ε, που έπληξε τη Μαδέρα και την Ατλαντική ακτή και ιδιαίτερα τη χώρα μου με δεκάδες νεκρών. Ε, και αυτή τη στιγμή θα ήθελα να επαναλάβω μια που έχω το λόγο ε, την αλληλεγγύη μας προς όλα τα θύματα και μετέβει ο συνάδελφός μου, ο αρμόδιος επίτροπος και εδώ θα πρέπει ε, ε, να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή πολλαπλασιάζονται οι θεομηνίες και έχουμε και άλλες ε, καταστροφές που δεν είναι πλέον φυσικές αλλά μπορούν να έχουν μεγάλες και σοβαρές συνέπειες για την ίδια τη ζωή ανδρών και γυναικών και για τη φύση και για την οικονομία. Ας πούμε, βιομηχανικές καταστροφές, πυρκαγιές, ναυάγια ή καταστροφές στη θάλασσα. Εδώ και χρόνια ασχολήθηκα με αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο από το 1999 ως φρέσκος επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική χρειάστηκε να απαντήσω σε έναν Έλληνα συνάδελφο ε, μετά του σεισμού στην Ελλάδα και τότε είχα προτείνει ε, τη δημιουργία πρώτων Ταμείου Αλληλεγγύης και στη συνέχεια μιας Ευρωπαϊκής Δύναμης Πολιτικής Προστασίας. Χρειάστηκε να ε, περιμένουμε το 2002 και τις μεγάλες πλημμύρες που έπληξαν η Γερμανία, Αυστρία και Σλοβακία και μέσα σε τρει μήνες με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το Ταμείο Λεγγύης το οποίο ε, θα ε, βοηθήσει και θα παρέμβει και στη Μαδέρα και στην ακτή του Ατλαντικού όπως και το έχει πράξει από το 2002. Η Ευρωπαϊκή Δύναμη προστασίας, Πολιτικής Προστασίας είναι θέμα της κυρίας Γεωργίευα και ε, της κυρίας ε, Άστον. Ελπίζω να μην χρειαστεί και νέα καταστροφή για να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για καταστροφές τύπου τσουνάμι ή αιτής. Το παρόν ερώτημα αφορά τις ασφάλειες. Γιατί δεν συνδέονται τα πάντα με δημόσια αγαθά ε, που δεν ασφαλίζονται, που εμπίπτουν στο Ταμείο Ελεγγύης. Νομίζω ότι χωράει πρόοδος εδώ ε, σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που καλύπτουν οι ασφάλειες. Ε, Λευκή βίβλος του 2009 για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή λέει ότι υπάρχει δημόσια στήριξη, ε, λήψη ιδιωτικής. Θα δώσουμε συνέχεια, θα δούμε πώς μπορούμε να ε, συμπληρώσουμε τα μέτρα αυτά με ιδιωτική ασφάλιση. Ζήτησα από τις υπηρεσίες μου να κάνουν μια συγκριτική αξιολόγηση, ένα benchmark και να μελετήσουν τι ισχύει στα διάφορα κράτη-μέλη και σε περιπτώσεις διασυνοριακού αντικτύπου και καταστροφών να έχουμε και ευρωπαϊκές ασφαλίσεις και όχι εθνικές. Γνωρίζω κύριε Κέλλη ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και ε, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους θα το μελετήσω με τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα κράτη-μέλη, τους εμπειρογνώμονες για να ανταλλάξουμε πρακτικές και να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, να τις ορίσουμε στο σωστό επίπεδο και ε, να προστατεύουμε καλύτερα τους πολίτες γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερες τέτοιες θεομηνίες. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δουλειά. Το screening, ε, μια καταγραφή λοιπόν των συστημάτων τι ισχύει σε κάθε χώρα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε κατά των θεομηνιών. Ευχαριστώ. Κύριε Κέλλη, μισό λεπτό για την συμπληρωματική σας ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Σαφώς μας ανησυχεί ιδιαίτερα η Μαδέρα και η Γαλλία και η χώρα μου. Ε, Ευτυχώ δεν είχαμε θύματα, αλλά ε, το ασφαλιστικό πρόβλημα φάνηκε πολύ γρήγορα. Οι περισσότεροι πολίτες δεν μπορούν να λάβουν ασφαλιστική κάλυψη αυτή τη στιγμή και σε μία πόλη ε, η οποία πριν από κάποια χρόνια είχε προβλήματα, η ασφάλιση ε, είχε πάρα πολλά... εξαπλασιάστηκε. Ε, Θα πρέπει ίσως να υπάρχουν και κυρώσεις κάποιες μορφής για αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ, ο κύριος Επίτροπος. Euh, directive, euh, Περιοδηγίας για τις πλημμύρες και κατά των πλημμυρών. Ανάγκες το 2007 έχουμε και ανακοινώσει τη επιτροπή από το 2009 για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών που είναι ανθρωπογενούς προέλευσης. Μιλάμε για οδηγίες πρόσφατες και ήδη έχουν αρχίσει να λειτουργούν ε, τα μέτρα που έχουμε προβλέψει. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον τα κάτι μέλη εφαρμόζουν ή όχι τα μέτρα που περιλαμβάνει η οδηγία για τις πλημμύρες. Το είδαμε στη Γαλλία και το έχουμε δει και στη χώρα σας. Υπήρξαν συνέπειες λόγω της ε, αύξησης των των περιοχών που οικοδομούνται, το πώς προστατεύονται από τις πλημμύρες οι ζώνες αυτές που οικοδομήθηκαν. Η Επιτροπή λοιπόν θα δει με προσοχή τι κάνουν τα κατημέλη και ιδίως τι δεν κάνουν και τι δεν υλοποιούν, θα δει κατά πόσο υπήρξαν παραβάσεις και αν εφαρμόζονται σωστά οι οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χίγκιν, συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιτροπό του για την απάντησή του. Όσον αφορά στο θέμα που έθεσε ο κύριος Κέλλη και την εφαρμογή της οδηγίας για τις πλημμύρες. Όπως ξέρετε, ε, θα πρέπει φέτος να με έχει μεταφορθεί και στα 27 κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέχει λίγο τις εθνικές αρχές για το κατά πόσον εφαρμόζεται. Το 1995 εγώ ήμουν υπουργό αρμόδιο για θέματα πλημμυρών στην Ιρλανδία και είπαμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη και κατασκευή κατοικιών και πλέον ε, αυτή τη στιγμή ζητούν αποζημιώσεις ε, άτομα τα οποία έχουν κατασκευάσει κατοικίε μετά το 1995. Επομένω, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο και να υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσει για τον οποιονδήποτε παραβιάζει αυτές τις, ε, ε τις υποχρεώσεις. Κύριε Μπαρνιέ, μήπως θα μπορούσαμε να ακούσουμε άλλη μια ερώτηση και να απαντήσετε και τις δύο. Κύριε Ζάμκα, έχετε το λόγο. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για ασφάλιση. Νομίζω ότι όταν έχουμε θεομηνίες, δύο πράγματα πρέπει να γίνονται και μάλιστα δύο πράγματα τα οποία πόρο απέχουν μεταξύ των. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως χρειαζόμαστε ένα κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει μια ενιαία κεντρική αρχή που θα μπορούσε να αντιμετωπίζει κρίσεις. Ε, φυσικές καταστροφές. Και επίσης, μήπως θα πρέπει να γίνει κάτι επιπλέον για να έχουμε καλύτερη πολιτική προστασία. Παραδείγματος χάρη δεν υπάρχουν αεροπλάνα. Χρειαζόμαστε μία κεντρική αρχή και χρειαζόμαστε και ε, δυνατότητες πολιτικής προστασίας. Ευχαριστώ, Επίτροπο. Δύο διαφορετικές ερωτήσεις εδώ. Καταρχάς, για το θέμα των πλημμυρών όπως Επίτροπος επιφορτισμένων τα θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών εδώ μου ζητήσατε να απαντήσω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Πώς, ε, τι κάνουμε με τις ασφάλειες, πώς αποζημιώνουμε τους ανθρώπους που είχαν υλικέ ζημιές σε προσωπικό επίπεδο. Θα κοιτάξω την πανοραμική αυτή εικόνα των διαφόρων ιδιωτικών ασφαλειών και τα προηγμένα συστήματα που υπάρχουν ε, για το τι γίνεται με χώρες που δεν έχουν ασφάλεια για την περίπτωση φυσικών καταστροφών λόγω χάρη ή τη Γαλλία που έχει σοβαρές αποζημιώσεις για τέτοιες φυσικές καταστροφές. Τώρα για τι πλημμύρες πιο συγκεκριμένα κύριε Βουλευτέ. Δεν είναι ακριβώ θέμα με το οποίο είμαι επιφαρτισμένο εγώ, με την ευθύνη του. Υπάρχει και ο Επίτροπο του Προβάλλοντο, ο οποίο θα μπορούσε να σα απαντήσει γραπτό, να σα πει πώ εφαρμόζονται ή όχι και, κατα... και εφαρμόζονται σωστά οι οδηγίε κατά των πλημμυρών. Όμω έχετε δίκιο. Το σημείο κλειδί εδώ είναι τι γίνεται με τι περιφερειακέ τοπικέ ε, πολιτικέ ε, στα θέματα τη κατασκευή κτηρίων, τη οικοδόμηση περιοχών. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα από τι Βρυξέλλε. Ο γενικό κανόνα είναι λογικό. Υπάρχουν ε, ζώνε και περιοχέ όπου δεν πρέπει να υπάρχει καμία κατασκευή κτηρίων. Μάλιστα, στη χώρα μου έχουν ψηφιστεί νόμοι ώστε συγκεκριμένα εργοστάσια να μεταφερθούν, να μετακινηθούν από ζώνε που πλήττονται συστηματικά από πλημμύρε. Και επίση να αποζημιωθούν κάτοικοι προκειμένου να μετακομίσουν πριν έχουμε καταστροφέ. Αυτό ήδη έγινε από το 1995. Αυτέ λοιπόν είναι ιδέε που θα τι εξετάσουμε από κοινού. Θα σκεφτούμε το τι γίνεται με τι ασφάλειε και θα προβούμε σε συγκεκριμένε προτάσει. Πάντως, ακόμη και αν αυτό είναι, μια, είναι αρμοδιότητα άλλου συναδέλφου, ξέρουμε ότι έχουν γίνει σχετικέ προτάσει από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει ήδη στηρίξει τι πρωτοβουλίε αυτέ ο πρόεδρο Μπαρόζο από το 2006 και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προστασία των Πολιτών θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και τη μορφή ενισχυμένη συνεργασία. Να κάνουμε μια προσέγγιση άντι δηλαδή να έχουμε κι άλλη συνεργασία, περαιτέρω συνεργασία των πολιτών. Με το τσουνάμι, με την τραγωδία τη ΑΕΤ είδαμε είδαμε τι συμβαίνει. Χρειάζεται σε πραγματικό χρόνο να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και βεβαίω να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή σε τέτοια θέματα. Εάν οι Ευρωπαίοι πολίτε μπορούν να ετοιμάσουν την απόκρισή του, την κατάλληλη απόκριση σε διαφορετικών ειδών φυσικέ καταστροφέ. Είναι άλλο πράγμα μια καταστροφή όπω το ναυάγιο της Έρικα, του Έρικα, ε, μια βιομηχανική καταστροφή, οι πυρκαγιέ στην Ελλάδα, οι πλημμύρε στη Γερμανία, το τσουνάμι ε, ή κάποιες τρομοκρατικέ απόπειρε όπως αυτή της ε, 11 Σεπτεμβρίου που ελπίζουμε να μην ε, λάβουν χώρα και στην Ευρώπη βεβαίως. Έχουμε τους συναδέλφους που εργάζονται και μοχθούν, θα έρθουν και προς εσάς και νομίζω θα ετοιμάσουν μια κοινή εύστοχη απάντηση για όλα αυτά τα θέματα. Άλλωστε και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να εργάζομαι με τη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Η επόμενη ερώτηση είναι προς τον κύριο Άντο. Σας περιμένουμε. And the question is number 30 by Mrs. Έχουμε την ερώτηση υπαριθμών 30 από την κυρία Τσικάου για τα ευρωπαϊκά μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Κατανοώ τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σε αυτή την ερώτηση για την ευημερία των Ευρωπαίων. Έχουμε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης της ένδειας. Όπως γνωρίζετε, το 2010 είναι το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της ένδειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για τα κοινωνικά προβλήματα και ελπίζουμε ότι φέτος θα είναι η κατάλληλη χρονιά ώστε να μην συζητήσουμε μόνο την ένδυα αλλά να αναλάβουμε και δεσμεύσεις για την καταπολέμησή της και να ανανεώσουμε την πολιτική δέσμευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μεταξύ όμως των κρατών μελών. Για να υπάρχει δυνατότητα ανενόησης αυτής της δέσμευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική και το 2020 έχει συμπεριλάβει ένα στόχο, πρωταρχικό στόχο για, τα, ε, για την καταπολέμηση της ένδυας και τα μαθήματα που μάθαμε από τα παρελθόν. Στόχος είναι να μειωθεί η ένδυα κατά το 1 τέταρτο, κατά 25% δηλαδή μέχρι το 2020. Θα πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας για όσους μπορούν να ε, συντηρήσουν τον εαυτό τους και αλληλεγγύη για όσους δεν μπορούν. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική για το 2020. Το να επιτύχουμε το στόχο λοιπόν τη καταπολέμηση τη ένδυα, θα πρέπει να έχουμε και μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία αποκαλείται πλατφόρμα κατά τη φτώχεια. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίηση και τη πρόσφατη πρωτοβουλία των μικροπιστώσεων. Οι δράσει που αναλαμβάνονται από τα κράτη-μέλη είναι εξίσου σημαντικέ. Βέβαια, θα πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι θέσει εργασία υψηλή ποιότητα είναι προσβάσιμε προ όλου. Η μείωση τη ένδυα θα πρέπει να πάει πέρα από τα θέματα τη απασχόληση διότι αναγνωρίζεται στην ανακοίνωση για το 2020 ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, αποτελεσματική, καλά σχεδιασμένη κοινωνική προστασία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ένδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τη χρηματοδότηση και την οργάνωση ε, συστημάτων κοινωνικής προστασίας με την υποστήριξη και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασικό στοιχείο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες πολιτικής και να διευκολύνουμε την αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη και γνώση. Υπάρχει ένα ενεργό πλαίσιο ε, ένταξης, ε, καταπολέμηση της παιδικής ένδυας και παρακολούθηση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσεως. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία των δύο Προεδριών του 2010, της Ισπανικής και της Βελγικής. Έχουν αναλυφθεί πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Το πρώτο στάδιο είναι η σύνδεση κορυφής των Ρωμά που συζητήθηκε μόλις πριν από λίγο εδώ ε, στην αίθουσα και υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός στόχος μείωση της ένδυας και κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας προετοιμάζουμε και μια πρωτοβουλία για τη μείωση της παιδικής φτώχειας. Δεν θα πρέπει βέβαια να συμμετάσχουν σε αυτό οι κυβερνήσεις μόνον. Χωρίς τη βοήθεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν θα μπορέσουμε να έχουμε επιτυχημένα προγράμματα. Είμαστε λοιπόν υπέρ ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα μείωση τη ένδυα. Αυτά είναι τα βασικά θέματα, τα οποία καλύπτουν βέβαια πολλέ κατευθύνσει ε, προ τι οποίε δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση τη ένδυα. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κύριε Τσικάου για συμπληρωματική ερώτηση. 30 δεύτερα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε ε, για την απάντησή σας. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά θα επιθυμούσα και θα μου άρεσε να συζητούμε λίγο και για τη διαδικασία αποβιομηχάνησης που βλέπουμε σε διάφορα κράτη-μέλη και είναι ένας από τους λόγους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που ζούμε. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική, κοινωνική, ευφυής, για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης. Ποια είναι λοιπόν τα μέτρα που προτίθεται να λάβετε για τη βιομηχανική πολιτική στο πρόγραμμα εργασία της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αυξηθούν και η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση στην Ένωση με εγγύηση για υψηλό βιωτικό επίπεδο και για αξιοπρεπέ βιωτικό επίπεδο για τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ, επίτροπο. Χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις απασχόλησης και καλύτερες και αυτές περιλαμβάνονται στη στρατηγική 2020 για την Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω την προσοχή και σε άλλες ε, πρωτοβουλίες πέρα από την ένδυα στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Θέσεις απασχόλησης ποιοτικέ και πολλές. Έχουμε τη νέα πρωτοβουλία Ναυαρχίδα ε, για τις θέσεις απασχόλησης και στο πυλώνα της αηφορίας ε, στο έγγραφο 2020 και υπάρχει και ιδιαίτερο κεφάλαιο για τη βιομηχανική πολιτική. Είναι θέμα κλειδί πραγματικά και πολύ καλή ερώτηση. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε δεν θα πρέπει να ασχολούνται μόνο με τις εταιρείες που εγκαταλείπουν την Ευρώπη, όπως είναι το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης που έρχεται να απαντήσει στην μετεγκατάσταση. Θα πρέπει να προλαμβάνουμε την απώλεια θέσεων απασχόλησης, τη φτώχεια ε, και τις δεξιότητες και θα ασχοληθούμε λοιπόν με τη βιομηχανική πολιτική για ε, αηφόρο οικονομία όπως αναφέρατε, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την ε, διατήρηση των εργοστασίων. Συμφωνώ απολύτως. Χωρίς συνολική προσέγγιση, χωρίς συνολική οικονομική πολιτική και πολιτική απασχόληση, δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε με επιτυχία την ένδυα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο επιπλέον ερωτήσεις. Ο κύριος Ρόμπερ Μάιερ και μετά ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακριβώ σε περιόδου οικονομική κρίση, ο κίνδυνο κατάχρηση των κοινωνικών θεμάτων είναι πολύ μεγάλο. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, υπάρχει πολύ μεγάλη κατάχρηση των κοινωνικών επιδομάτων και τις ελάχιστες ε, συντάξεις ε, από τα νέα κράτη-μέλη ζητούν αντισταθμίσεις οι πολίτες πολύ περισσότερες από την ίδια τους τη σύνταξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει, θα δώσει στα κράτη-μέλη μονομένα εργαλεία για να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ε, της ε, κατάχρησης των επιδομάτων και των συντάξεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χουντή, παρακαλώ. 30 δεύτερα. Συγγνώμη, να ρωτήσει πρώτα ο κύριος Χουντή για να απαντήσετε. Κύριε Επίτροπε, στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω από τα όρια τη φτώχεια είναι πάνω από 20%. Από αυτού, σε συνθήκες φτώχειας 34% είναι άνεργοι και υπάρχει και ένα ποσοστό 14% εργαζομένων φτωχών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το πρόβλημα της φτώχειας που περιέγραψε η συνάδελφος με την ερώτηση σε σχέση με την Ευρώπη και τα στοιχεία που σας έδωσα για την Ελλάδα κατά τη γνώμη μου οφείλονται στην αποτυχία του νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου που προωθούσε η συνθήκη της Λισαβόνα και το επαναφέρει το κείμενο της στρατηγικής 2020. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα αυξανόμενα ποσοστά φτώχεια με αποσπασματικέ πολιτικέ που έχουν και στοιχεία φιλανθρωπίας ή χρειάζεται μια άλλη οικονομική πολιτική που να έχει στο επίκεντρό τη την πλήρη απασχόληση και επομένω πρέπει να ξαναδείτε το κείμενο τη ευρωπαϊκή στρατηγική. 2020. Ευχαριστώ. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω με τη δεύτερη ερώτηση, αν δεν σας πειράζει. Είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα πιο σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον. Στην προηγούμενη απάντησή μου αναφέρθηκα στη σημασία μιας πλήρους οικονομικής πολιτικής, ώστε να έχουμε ένα πιο σταθερό περιβάλλον. Πράγματι λοιπόν, αυτό που αναφέρατε εσείς ως νεοφιλελευθεριστική τάση των τελευταίων δεκαετιών θα πρέπει να αναθεωρηθεί και στην Ευρώπη του 2020 διαπιστώνεται κάποιες ε, μια σειρά από πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να σταθώ στο κεφάλαιο του χρηματοοικονομικού κανονισμού που περιλαμβάνει αρκετά σοβαρές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς και προκύπτει ακριβώς επειδή υπάρχει πρόθεση να έχουμε ένα σταθερότερο μακροοικονομικό περιβάλλον, γεγονός που θα μειώσει τις πιέσεις των φορολογικών συστημάτων τα οποία στόχο έχουν να ε, υποστηρίξουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και τις ε, ε, κοινωνικές πολιτικές. Όσον αφορά τώρα την κατάχρηση και το κατά πόσον είναι αποτελεσματικά τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, η κρίση αποτελεί μια δοκιμή υπό αυτήν την έννοια. Αυτό που μπορεί λοιπόν να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο ανοιχτού συντονισμού και τι δυνατότητε παρακολούθησης, εποπτείας και εκθέσεων για να παρακολουθεί καλύτερα τα μέτρα κοινωνική προστασία που λαμβάνονται η πρόκληση εν καιρό κρίσης ε, που αναφέρθηκε, ε, αλλά και για το επόμενο χρονικό διάστημα, ε, είναι ότι τα κράτη-μέλη θα χρειαστούν παγίωση από φορολογικής πλευράς. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να εξεύρουμε περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση της ένδυας. Μας είναι λοιπόν χρήσιμο να ανταλλάσσουμε εμπειρίες για να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα συστήματά μας και πώς μπορούμε να στοχεύσουμε στις ευάλωτες ομάδες με καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Να περάσουμε τώρα στην ερώτηση παριθμών 31. Η κυρία Βασιλείου θα απαντήσει. Η ερώτηση είναι από τον κύριο για την αξιολόγηση του προγράμματος Culture 2007-2013. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη, όπως ε, αναφέρει ο βουλευτής ε, Παπα-Νικολάου, στόχος του προγράμματος «Πολιτισμός» είναι ο εμπλουτισμός της πολιτιστικής εμπειρίας των Ευρωπαίων πολιτών με την προβολή της κοινή μα πολιτιστικής κληρονομιάς. η επιτροπή προωθεί την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των δημιουργών των πολιτιστικών φορέων και των θεσμών των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με σκοπό την ενθάρρυνση της διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής υπηκότητας. το πρόγραμμα πολιτισμός στοχεύει ειδικότερα στην προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών φορέων στην ενθάρρυνση της διακρατικής κυκλοφορία των καλλιτεχνών και πολιτιστικών έργων και προϊόντων και στη στήριξη του διαπολιτισμικού διαλόγου. ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2009 στο πλαίσιο του προγράμματο Πολιτισμό, υποβλήθηκαν 749 αιτήσει και επελέγησαν 256 σχέδια για χρηματοδότηση από τα οποία τα 127 είχαν ω κύριο στόχο την κινητικότητα των πολιτιστικών φορέων. σύμφωνα με τη νομική βάση απαιτείται τακτική εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση του προγράμματος. τον ιούλιο του 2009 η επιτροπή κάλεσε ανεξάρτητο ανάδοχο να αξιολογήσει τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής του προγράμματος πολιτισμός Πολιτισμός χιλιάδες και ειδικότερα τη συνάφεια των στόχων τα πρώτα αποτελέσματα και τον αρχικό αντίκτυπο του προγράμματος. ο ανάδοχος πραγματοποιεί την αξιολόγηση με βάση τα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των σχεδίων τις πρόσφατες μεμονωμένες αξιολογήσεις τις έρευνες και συνεντεύξεις με τους δικαιούχους σχεδίων και τους ενδιαφερόμενους πολιτιστικούς φορείς. η τελική έκθεση του θα υποβληθεί το δεύτερο εξάμεινο αυτού του χρόνου. σε αυτή τη βάση η επιτροπή θα συντάξει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος και θα την υποβάλει στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το αργότερο μέχρι τις 31 δεκεμβρίου του. 2010. Παρακαλώ σημειώστε, κυρίες και κύριοι βουλευτές ότι το πρόγραμμα δεν στοχεύει πρώτιστα στις εθνικές αρχές αλλά στους πολιτιστικούς φορείς. Η συμμετοχή των πολιτιστικών φορέων σε σχέδια είναι σχετικά ομοιόμορφα κατανεμημένη στα κράτη-μέλη. Οι εθνικές αρχές συμμετέχουν σε ομάδες εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση της πολιτικής ανάπτυξης του προγράμματος. μετά από δύο γύρους πιλωτικών σχεδίων για την κινητικότητα των καλλιτεχνών που εγκαινιάστηκαν ε, από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για το 2008 και 2009 και λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις που ήδη διεξάγονται στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού η επιτροπή σε αυτό το στάδιο αξιολογεί την πρόοδο που έγινε μέχρι στιγμής και εξετάζει τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής του τρέχοντος προγράμματος. αργότερα εντός του έτους η επιτροπή θα αρχίσει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για να προετοιμαστεί το έδαφος για το νέο πρόγραμμα πολιτισμός για το έτος δύο και μετέπειτα. ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση, ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας κυρία Επίτροπε. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που είστε μαζί μας σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή δύναμη. Ε, πράγματι είναι καθοριστική η ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών στα πολιτιστικά στοιχεία που έχουν σημασία για την ευρώπη και αποτελούν σημεία αναφορά του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των κοινών αξιών μας και νομίζω το σημείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα το τελευταίο χρονικό διάστημα και για την ελλάδα και επιτρέψτε μου έτσι να προχωρήσω λίγο τη συζήτηση υπό το βάρο τη χρησιμοποίηση πολιτιστικών μνημείων για άσχετου με τον πολιτισμό λόγου, προκειμένου να ειρωνευτούν τη χώρα μου. αναφέρομαι στο δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού focus με την παραποίηση της αφροδίτης της μήλου αναφέρομαι στα διαδικτυακά δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την ακρόπολη ως ένα ερείπιο. υπό το φόβο λοιπόν μήπως πλέον αυτή η πρακτική δεν αποτελέσει εξαίρεση ερωτώ εσάς αξιότιμη κυρία επίτροπε αν καταδικάζετε αυτές τις πρακτικές και αν στα πλαίσια του προγράμματος που συζητάμε αλλά και όχι μόνο αν η επιτροπή σχεδιάζει την ανάληψη μιας πιο αποφασιστικής πιο επιθετικής επιτρέψτε μου να πω πολιτικής για την προώθηση του πολιτισμικού Συγγνώμη, μισό λεπτό είναι για την επερώτηση και ήδη έχουμε πολλή καθυστέρηση και πολλές ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Βασιλείου. Να μου επιτρέψετε να μην ε, εγώ ε, αυτή τη στιγμή παρατηρήσεις για δημοσιεύματα τα οποία δημοσιεύονται σε διάφορα έντυπα διότι πραγματικά εάν αρχίζαμε να ε, απαντούμε σε δημοσιεύματα αυτού του είδους νομίζω δεν θα καταλήγαμε πουθενά. Ε, εκείνο το οποίο λέω είναι ότι πολιτιστικά μνημεία όπως η Ακρόπολη και άλλα μνημεία της ελλάδος και άλλων χωρών μελών αποτελούν έναν ε, ε, θέλετε πηγή έμπνευσης και πολιτιστικής διαπολιτισμικής ε, αν πλούτου και ακριβώς σήμερα η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει υιοθετήσει ένα νέο σύστημα για σήμανση των μεγάλων ε, πολιτιστικών μνημείων της ευρωπαϊκής ένωσης μεταξύ των οποίων είναι και ο παρθενώνας και η ακρόπολης. αυτό νομίζω μιλά από μόνο του όσον αφορά το πώς σκέφτεται η ευρώπη για αυτά τα μνημεία. Ε, Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ερώτηση αυτή. Η επόμενη είναι η 32 από τον κύριο Έλβολτ για τους ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενίσχυση και χρηματοδότησή τους. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Αναγνωρίζουμε πλήρως τους ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό εστιάζει στην ε, πτυχή της κοινωνίας που ασχολείται με τον αθλητισμό και ε, αναφέρει μια σειρά από δράσεις που μπορούν να αυξήσουν την ε, σωματική δραστηριότητα, τη σημασία του αθλητισμού ε, που μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη σε ομαδικά αθλήματα και όλες αυτές οι δράσεις εφαρμόστηκαν ή είναι στη φάση εφαρμογής τους στο άρθρο 165 ενισχύεται με τη νέα συνθήκη ε, ο αθλητισμός και τονίζεται πόσο σημαντικός είναι και πόσο κοινωνική και εκπαιδευτική λειτουργία έχει και βασίζεται σε δομές ε, που προάγουν τον αθλητισμό. Αυτό μας δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ε, προαγωγή του αθλητισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ευρωπαϊκές δράσεις και προάγεται η ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει πρωτοβουλίε για την εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα στον τομέα του αθλητισμού στη διάρκεια του τρέχοντο έτου και θα λάβουμε υπόψη και την ανάγκη να ενισχύσουμε του ερασιτεχνικού ε, αθλητικού ε, συλλόγου. Ο αξιότιμος Ευρωβουλευτής σωστά επισημαίνει ότι αυτές οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν σχηματικές προκλήσεις ε, στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Μελέτη για τους εσωτερικούς φραγμούς της αγοράς ε, για τον αθλητισμό που αναφέρθηκε στην ε, Λευκή Βίβλο και εστιάζει και στη χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών σου λόγων, αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις. Η μελέτη στόχο έχει να καθορίσει ποιες είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης και να εντοπίσει μοντέλα χρηματοδότησης ε, στα διάφορα κράτη-μέλη και μάλιστα για διάφορα αθλήματα προκειμένου να αναλύσει το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και τις εθνικές πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στην χρηματοδότηση του αθλητισμού. Τέλος, η μελέτη θα πρέπει να επισημάνει κάποια αποτελεσματικά επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία ίσως θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικέ προκλήσεις όπως για παράδειγμα τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον κρατικό προϋπολογισμό και στις χορηγίες καθώς επίσης και να εντοπίσει τα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τους ερασιτεχνικούς ε, αθλητικούς συλλόγους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαβολεύσεις για τη χρηματοδότηση στα αεραστεχνικά σωματεία, τα οποία αναφέρει εδώ ο αξιότιμος Ευρωβουλευτής, συζητήθηκαν στα πλαίσια αυτής της μελέτης. Τα αρχικά αποτελέσματα καταδεικνύουν βάσει των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν σε ε, φόρουμ ενδιαφερομένων ε, ότι πρέπει να γίνουν στοιχεία για την εσωτερική αγορά και ο χορηγός στις 16 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες παρουσίασε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της διάσκεψης θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Έλβορτ για την επερώτηση για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την απάντησή της και θα καλωσορίσω τη δεσμεύση αυτή για να στηρίξουν το επίπεδο χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων. Λόγω τη ε, κύρωση τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα, νομίζω ότι έχουμε πλέον αρμοδιότητα και στον τομέα των αθλητικών και υπάρχει και ανάλογο κονδύλιο στον προπολογισμό. Το ερώτημα στην Επιτροπή είναι πώ σκοπεύει να σχηματίσει το πρόγραμμα αθλητισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση που περιμένουμε από την Επιτροπή για το θέμα αυτό, πότε προβλέπεται να ετοιμαστεί. Έχετε το λόγο. Η ανακοίνωση για τον αθλητισμό και την προογή του ε, θα κατατεθεί το καλοκαίρι πριν τις ελληνές διακοπές ε, για να θέσει το πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας και ε, μιας νέας ατζέντα για τον αθλητισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα σχέδιο απόφασης για ένα διετές πρόγραμμα για τον αθλητισμό 2012-2013. Βεβαίως, στο μεταξύ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, Έχουμε δράσει για τον αθλητισμό από το 2009, 2010, 2011. Συνεχίζεται και εστιάζει ακριβώς ε, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, στην κοινωνική διάσταση του αθλητισμού και Εγκρίθηκαν οι δράσεις αυτές ήδη από το 2009 και όπως γνωρίζετε φέτος εφαρμόζονται. Αυτό τον καιρό ε, ετοιμαζόμαστε να εγκρίνουμε τη δράση για το 2010. Σε μερικούς μήνες θα έχει ολοκληρωθεί πιστεύω. Και σύμφωνα με τον προεπολογισμό που έχουμε, διότι όπως επίσης γνωρίζετε πολύ καλά, ο προπολογισμό για το 2010 έχει περικοπεί από τα 6 στα 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, σύμφωνα με τον προπολογισμό που έχουμε και για το 2011, προβλέπουμε νέες δράσεις και νέο υλικό ε, να δοκιμάσουμε για να ε, διατυπώσουμε το πρόγραμμά μας για το 2012-2013. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόης έχει συμπροματική ερώτηση για μισό λεπτό. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος για όσα μας αναπτύξατε για την νέα στρατηγική για τον αθλητισμό. Θα ήθελα όμως να αναφέρω και κάτι ακόμη που συζητιέται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Πολιτισμού μας ε, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Νέες αρμοδιότητες, καθοριστικής σημασίας μάλιστα, όπως η γνώση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον αθλητισμό. Γνώση για τον αθλητισμό λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει έμφαση σε τέτοια στοιχεία όπως ο αθλητισμός και η γνώση περί αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προαγωγή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι σημαντικά όλα αυτά για την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλώ βέβαια για τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, ε, θεωρώ επίσης πολύ σημαντικά θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, και συνεργασία για να σφυριλατηθεί η κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητά μας. Βεβαίως θα ληφθούν όλα αυτά υπόψη όταν θα κάνουμε ένα μονιμότερο πρόγραμμα για τον αθλητισμό. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Ολοκληρώνεται εδώ ε, γύρω των ερωτήσεων που απευθύνονται σε εσά και ακολουθούν οι ερωτήσει προς τον κύριο Κάλλας. Παρακαλώ. And, ε, The first of the Η πρώτη ερώτηση είναι η 33 από τον Jim Higgins για το θάνατο από τροχαία ατυχήματα. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στα πλαίσια του τρίτου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τα οδικά ατυχήματα το 2010, είχαμε μια σειρά από δράσεις για να καταπολεμήσουμε την ε, ε, ταχύτητα, την ε, οδήγηση υπό τον επίρρεια μέθης ναρκωτικών και την ανεπαρκή υποδομή του οδικού δικτύου και συμμετείχε φυσικά και το Κοινοβούλιο βάσει διαδικασία συναπόφεσης. Βέβαια χρειαζόμαστε περαιτέρω μέτρα. αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την ευρωπαϊκή πολιτική για τα οδικά δυστυχήματα. Ε, μας ενδιαφέρει κυρίως ε, η ταχύτητα, η οδηγία επί των μέθης ναρκωτικών και οι υποδομές διότι φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, δεν ε, κατανοούν γιατί δεν τιμωρούνται όσοι προκαλούν ατυχήματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ε, μία οδηγία για την αντιμετώπιση των διαμεθοριακών ε, προβλημάτων όπως ε, ακριβώς ζήτησε το Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει την πρόταση αυτή και πέρα από τις κυρώσεις μας ενδιαφέρουν και η κατάλληλη παιδεία και η ευαισθητοποίηση σε θέματα αυτά. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένε δράσεις για την κατανάλωση αλκοόλ και την ταχύτητα ε, και καθώς και αυστηρότερες απαιτήσεις ε, για τους ε, οδηγούς που οδηγούν υπό την επίρρεια μέθης. Έχουμε και συνεχιζόμενα ερευνητικά προγράμματα για να μας δώσουν νέες ιδέες για την αντιμετώπιση του θέματος. Όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχει υιοθετηθεί νομοθεσία για την ασφάλεια και τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου και περιμένουμε τώρα την εφαρμογή από πλευράς κρατών μελών. Η οδική ασφάλεια και οι κατάλληλες υποδομές ε, δεν περιορίζονται μόνο στους βασικούς 10 ε, οδικούς άξονες, ε, διότι πάρα πολλά ατυχήματα συμβαίνουν και σε υπαίθριους αυτοκινητοδρόμους. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να προεκτείνουμε την παρούσα οδηγία για την ασφάλεια ε, στους δρόμους ε, και στους ε, υπαίθριους αυτοκινητοδρόμους. Θα πρέπει λοιπόν, επαρχιακούς αυτοκινητοδρόμους, θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες απαιτήσει ασφαλείας και ε, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτό είναι κοινή ευθύνη μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, κρατών μελών, περιφερειακών ε, φορέων και φυσικά και των πολιτών. Για να έχουμε λύσει, θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στου δρόμου και η επόμενη στρατηγική για την οδική ασφάλεια θα προτείνει μια σειρά από δράσεις που θα βασίζονται σε αυτή την αρχή. Στόχο είναι να υπάρχει ένα κοινό χώρο οδική ασφάλεια ο οποίος ε, θα αποτελεί και τμήμα του ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και όλοι οι πολίτες θα απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ασφαλείας ε, στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χίγκες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο. Ακούγοντας το καταλαβαίνει κανείς ότι έχει κάνει πολλά ε, για την καταπολέμηση της υπερβολικής ταχύτητας και του ινοπνεύματος, ε, αλλά για τα ναρκωτικά ούτε έρευνα δεν κάνετε. Είναι μεγάλο το πρόβλημα όταν κανένας οδηγεί υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ. Κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους 10.000 Ευρωπαίοι σε τροχιά δυστυχήματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ναρκωτικών. Είναι ε, μεγάλο αίτιο, ευθύνεται για πολλά ε, δυστυχήματα και θανατηφόρα τροχέα. Και θα ήθελα να συστήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πολλά περισσότερα για τα ναρκωτικά συγκεκριμένα. Κατανοώ και καλωσορίζω αυτά που κάνετε, αλλά χρειάζονται περισσότερα. Ευχαριστώ. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ παρά να συμμεριστώ τις ανησυχίες σας. Όμως, το πρόβλημα είναι, όπως ξέρετε, όταν χρειάζονται προηγμένα τεχνολογικά μέσα για να το εντοπίσει κανείς τους οδηγούς που βρίσκονται υπό την επίρρεια του αλκοόλ, μέθης δηλαδή. Άλλωστε η επίρρεια των ναρκωτικών είναι πολύ πιο δύσκολο να ανοιχνευτεί. Οπότε πώς να κάνουμε έρευνα και πώς να έχουμε και στα χέρια μας αμέσως την απαραίτητη τεχνολογία. Διότι αυτή τη στιγμή η πρώτη παρατήρηση που μπορούν να κάνουν οι αστυνομικοί όταν υποβάλλουν σε έλεγχο τους οδηγούς δεν μπορούν να το τα πάντα. Χρειάζονται σίγουρα περισσότερα. Μάλιστα. Δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις έχω. Ο κανόνας είναι στην ώρα των ερωτήσεων ότι μόνο δύο επερωτήσεις επιτρέπονται ερώτηση. Και θα πρέπει να διατηρηθεί και κάποια ισορροπία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Μπαλσίτη και ο κύριο Χουντή. Πρώτος ο κύριο Μπαλσίτη. Μισό λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας και την απάντησή σας. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τι λέτε για τα κινητά τηλέφωνα κατά την οδήγηση και η χρήση των κινητών δεν είναι ένα από τα αίτια θανατηφόρων δυστυχημάτων στους δρόμους μας. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αποσπάται η προσοχή των οδηγών όταν μιλούν στο τηλέφωνο. Σαν να έχουν πάρει ναρκωτικά ή να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και άλλος παράγοντας κινδύνου είναι όταν οδηγεί κανείς τη νύχτα. Ε, βαριά ε, φορτηγά δημόσιας χρήσης σε κακούς δρόμους. Λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε. Μήπως θα πρέπει να περάσει το σιδηρόδρομο η μεταφορά των εμπορευμάτων, αντί να είναι οδική. Ο κύριος Χοντής. Το θέμα που συζητάμε είναι πάρα πολύ σοβαρό, το θέμα που έθιξε ο κύριος συνάδελφος με την ερώτησή του. Αυτό που λέμε τροχαία ατυχήματα, κατά τη γνώμη μου, είναι συγκρούσεις που οφείλονται σε πολλές αιτίες και είναι πράγματι η αιτία πολλών θανάτων στην Ευρώπη θέλω να σα ρωτήσω δύο λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα. πρώτον επειδή οι περισσότερε αυτέ συγκρούσει γίνονται στι πόλει με περισσότερα θύματα του πεζού και του ποδηλάτε τι πρωτοβουλίε βλέπετε ότι πρέπει να αναπτυχθούν τόσο ώστε να πάμε στη λογική αυτό που λέμε vision zero δηλαδή να μην έχουμε θύματα στι πόλει να προσέχουμε ιδιαίτερα τα σχολεία του ποδηλατόδρομου και ούτω καθεξής. και η δεύτερη ερώτηση είναι τι προτίθεστε να κάνετε ούτω ώστε να απονέμεται δικαιοσύνη υπέρ των θυμάτων και των συγγενών στο πλαίσιο τη λογική ούτω ώστε με αυτή τη λογική να πετύχουμε και την πρόληψη των ατυχημάτων. Κύριε <clears throat> έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά η αλλαγή των ε, μέσων μεταφοράς όπως ε, καλείται, το να προτιμούμε για παράδειγμα τους σιδηροδρόμους, είναι σαφής προτίμηση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αποτελούσε και επιθυμία μας, διακαή μας επιθυμία τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα βοτιγλιαρίσματα πώς μπορούμε να τα καταργήσουμε τα οποία δεν μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πλεονεκτήματα των σιδηροδρόμων. Φαντάζομαι ότι στη διάρκεια της θητείας ε, της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Το μόνο που μπορώ να πω για τη χρήση κινητών τηλεφώνων είναι ότι τουλάχιστον σε κάποιες χώρες και στη δική μου τη χώρα απαγορεύεται η χρήση ε, κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Οι δράσεις τώρα για την αντιμετώπιση των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων, η Επιτροπή είχε ένα φιλόδοξο στόχο να μειώσει τον αριθμό των ε, θυμάτων κατά 50%. Δεν επετέχθη βέβαια, αλλά υπήρξε ουσιαστική μείωση της θνησιμότητας και αυτό ήταν ε, αποτέλεσμα και της δουλειάς των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων αλλά και των κρατών μελών. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, η μείωση των ε, θυμάτων ήταν αξιοσημείωτη την τελευταία δεκαετία. Μειώθηκε κατά τρεις φορές. Ελπίζω να μειωθεί σημαντικά και για το μέλλον. Σίγουρα δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε στα μηδενικά ε, θύματα, αλλά ε, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον αριθμό των θυμάτων. Είναι περίπλοκο το ζήτημα. Έχουμε αντιμετώπιση ε, της οδηγίας υποκατάσταση μέθης, καλύτερη παιδεία και μία σειρά από άλλα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι κοινή από τον Ιβο Μπέλετ και τη Φρίντα Μπρίπερ σε ερωτήσει 34 34 και 35 για το σιδηροδρομικό ατύχημα στο Μπούλτζικεν και το ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας και τα αίτια του τραγικού σιδηροδρομικού ατυχήματος στις 15 Φεβρουαρίου. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη. Το σιδηροδρομικό ατύχημα στο Μπούλτζικεν τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου ήταν φυσικά μια τραγωδία. Και ε, στη συνέχεια ε, αυτού του ατυχήματος ε, μπορούν να τεθούν πολλά ερωτήματα τεχνικής και πολιτικής φύσεων. Έχει ξεκινήσει μία έρευνα για τους τεχνικούς λόγους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για θέματα ασφάλειας και είναι αρμοδιότητα της βελγικής κυβέρνησης να ερευνήσει το θέμα και φυσικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιδηροδρόμων θα πρέπει να συμμετέχει. Ο η βελγική πλευρά ξεκίνησε την έρευνα λίγες ώρες μετά το δυστύχημα. Δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί τα αίτια και επομένως είναι ε, αδόκιμο προς το παρόν να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Κάθε φορά που υπάρχει σιδηροδρομικό ατύχημα υπάρχουν ε, παρατηρήσεις ε, για την, για την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι το άνοιγμα της αγοράς κυρίως και του σιδηροδρομικού τομέα στον ανταγωνισμό και στον καθορισμό απαιτήσεων για να υπάρχουν ε, ε, ξεχωριστές διαχειριστικές αρχές και διαχείριση των σιδηροδρόμων ε, μας ε, ενδιέφερε ε, ιδιαίτερος εξ αρχής. Παρακολουθούσαμε το άνοιγμα του τομέα των σιδηροδρόμων ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και να μην υπάρχει καμία τέτοια επίπτωση ε, Γι' αυτό ακριβώς και δεν θεωρώ ότι υπάρχει σχέση ε, μεταξύ του δυστυχήματος αυτού και ε, το ερώτημα που στείλαμε στην βελγική κυβέρνηση πριν από κάποια χρόνια. Οποιαδήποτε ερώτηση συνδέει την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους με την ε, απελευθέρωση της αγοράς, κατ' εμέ δεν έχει λόγο ύπαρξης. Έχουμε πάνω από 20 διαφορετικά εθνικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την ε, ε, ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Το γεγονός ότι αυτά τα συστήματα είναι ασύμβατα προκαλεί μεγάλα προβλήματα διότι θα πρέπει να αλλάξουν οι σιδηρόδρομοι στα σύνορα και ορισμένες φορές ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διπλά συστήματα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να υπάρχει νέα σύστημα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο έχει σχεδιαστεί, έχει αναπτυχθεί και αυτή τη στιγμή είναι στη φάση της υλοποίησής του. Ε, το σύστημα είναι γνωστό ως ERTMS, ε, Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας των Σιδηροδρόμων. Επίσης, αναπτύχθηκαν κάποια συστήματα στη διάρκεια της δεκαετίας του 80, αλλά η πλήρης εφαρμογή του είναι μια μακροπρόθεσμα διαδικασία. Στις περισσότερες χώρες που υπάρχει αυτό το σύστημα, Υπάρχουν αρκετά ε, δίκτυα ε, τα οποία είναι εξοπλισμένα και ο εξοπλισμός ε, διέρχεται περίπου 20 χρόνια. Έχουν δημιουργηθεί προδιαγραφές από το 2000 και έχουμε και κάποια πιλωτικά προγράμματα μεταξύ 2000-2005. Από το 2005 και λοιπά υπάρχουν αρκετές, και μετά συγγνώμη, υπάρχουν αρκετές γραμμές οι οποίες είναι εξοπλισμένες με το ERTMS. Υπάρχουν επίσης και προγράμματα ανεξελίξης σε όλα τα κράτη-μέλη. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, η γραμμή Λιέγη-Άχεν είναι εξοπλισμένη με το σύστημα και οι σειρμοί Intercity ε, διαθέτουν το σύστημα αυτό. Το σύστημα αυτό ε, θα συνεπάρχει κατά πάσα πιθανότητα με τα εθνικά συστήματα για ένα διάστημα 20 ετών ε, Κάποια κράτη-μέλη θα χρησιμοποιούν το εθνικό του σύστημα και κάποια άλλοι θα χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό σύστημα. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι το ισπανικό και το ιταλικό σύστημα ήδη διαθέτουν ε, το ERTMS, ε, το Λουξεμβούργο επίσης, αλλά σε, κάποια, σε 15 κράτη-μέλη έχουμε μόνο πιλωτικές γραμμές. Θα πρέπει επίσης ε, να αναφέρουμε ότι τα συστήματα αυτόματης προστασίας είναι μόνο ένα από τα μέτρα. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης κατάλληλη κατάρτιση, ε, καλύτερη προστασία στους, ε, στις διασταυρώσεις ε, και καθώς και άλλα μέτρα για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη κάλυψη. Αν λάβουμε υπόψη τους δείκτες ασφαλείας, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι σιδηρόδρομοι είναι σε γενικές γραμμές αρκετά ασφαλείς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Μπελέτ και μετά η κυρία ε, Μπρέπουλς για τις ερωτήσεις τους για να απαντήσετε στη συνέχεια. Μισό λεπτό ο κύριος Ιβο Μπελέτ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ποιο δίδαγμα θα πρέπει να βγάλουμε από αυτό το δράμα, τη τραγωδία. Θα γίνει ειδική επιτροπή, ξέρετε, στο Βελγικό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να καταλήξουν οι βελγικές αρχές. Ερώτηση τι λέτε για τα κοινωνικά στοιχεία και το φόρτο εργασίας που έχουν οι μηχανοδηγοί και γενικά το προσωπικό, ε, το σιδηροδρομικό. Αυτό δεν θα το κοιτάξετε. Μήπως χρειάζεται ε, ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση γιατί θα αυξηθεί και ο ανταγωνισμός τα επόμενα χρόνια στον τομέα της μεταφοράς επιβατών. Η κυρία Μπρέπουλς, παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ θερμά τον Επίτροπο για την απάντηση που έδωσε. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, απάντηση. Τη δική μου δεν την απάντησε όμως. για την αιτηρογημένη γνώμη που έστειλε το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Βέλγιο. Το 2009 επίσης διαπίστωσε ότι η Infrabel ε, δεν είναι ανεξάρτητη από τους βελγικούς σιδηροδρόμους. Πόσο χρόνο δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων του Βελγίου για να κάνει τις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις και προσαρμογές. Έχετε το λόγο παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Πρώτον, για τους διαχειριστές ε, του δικτύου και τα κοινωνικά ζητήματα. Βεβαίως, Μπορεί κανείς να κάνει μελέτες και αναλύσεις της κατάστασης, αλλά όταν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και πολύ πυκνή κυκλοφορία, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά και αυτό της πίεσης και το, κοινωνικό θέμα. Υπάρχουν ήδη πολλοί κανονισμοί, ξέρετε, που αφορούν ε, τους χειριστές αεροσκαφών ή ε, την οδηγία για τους χρόνους οδήγησης στις οδικές μεταφορές. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν ε, θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος για το πόσες ώρες εργάζονται οι μηχανοδηγοί ε, όπως και οι υπόλοιποι οδηγοί άλλων οχημάτων. Βεβαίω και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά πάντα υπάρχει και εθνική νομοθεσία, ξέρετε. Και κατά πρώτο λόγο αυτά είναι ζητήματα εθνικής νομοθεσίας. Βεβαίω είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008, σας είπα και προηγουμένως, απίφθινε στο Βέλγιο αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία επέκρινε επισήμως ε, την ε, έλλειψη εγγύσεων ε, ανεξαρτησίας του διαχειριστή σε ό,τι αφορά το τροχαίο υλικό και το φορτίο. Απάντησαν οι βελγικές αρχές και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλύουν την απάντηση αυτή. Βεβαίω είναι τραγωδία το δυστύχημα αυτό που συνέβη το σιδηροδρομικό και θα έπρεπε να είχε αποφευθεί αλλά ποτέ στον κόσμο δεν υπάρχει απόλυτη μηδενική ε, απόλυτη ασφάλεια συγγνώμη, και, και μηδενικά δυστυχήματα. Και ανεξάρτητα από τα αιτία είναι πάντα τραγική συγκυρία και ε, πολλά τα αίτια και ο ανθρώπινος παράγοντας. Από το 19ο αιώνα ξέρουμε ότι το κόκκινο φανάρι σημαίνει stop και πρέπει να σταματήσεις. Βέβαια δεν είναι απλή απάντηση σε αυτό το δυστύχημα γιατί συνέβη. Ευχαριστώ. Now, Mr. Boris, a supplementary half a minute. Ε, μισό λεπτό, συμπληρωματική ερώτηση ο κύριος Μπόρις. Ε, επίτροπε, αυτή την τραγωδία πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως αφορμή για να αντλήσουμε διδάγματα. Δεν ξέρουμε ακόμα αν το σφάλμα ήταν ανθρώπινο, τεχνικό ή σφάλμα του δικτύου. Η Επιτροπή πότε πιστεύει ότι η ERTMS μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται, το σύστημα αυτό. στην σιδηροδρομική, στη δίκτυα για εμπορεύματα και επιβάτε. Δεν πιστεύω ότι να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγηση τη ποιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Το σχέδιο είναι το σύστημα ERTMS να αρχίσει να χρησιμοποιείται ως βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο για όλη την Ευρώπη πριν το 2015. Ελπίζουμε ότι ως τότε αυτό το σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιείται ήδη. Όμως δεν σημαίνει ότι και οι περιφερειακές και τοπικές γραμμές θα έχουν εξοπλιστεί με αυτή την προηγμένη τεχνολογική με αυτό το προηγμένο τεχνολογικό δίκτυο τόσο γρήγορα. Είναι όμως ένας από τους στόχους που έχουμε και είναι και μια βέβαια δαπανηρή η διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα για την Αξιολόγηση και τη Μέτρηση της Ποιότητας είναι πολύ ωραία ιδέα σας Και όταν εξέφρασα την ιδέα να αναπτύξουμε τις μεταφορές συνολικά για την Ευρώπη, για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών, αυτό υπονοεί ότι θα πρέπει να ενοποιήσουμε και να ευθυγραμμίσουμε τις απαιτήσει ποιότητας. Θα πρέπει να έχουμε το, όσο πιο ψηλά γίνεται τον πύχη για την ποιότητα εκεί. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση του κυρίου Βρόσοβιτς για την αλλαγή της ώρας. Έχετε το λόγο κύριε Επιτροπέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, έχουμε οδηγία από το 2001 τον Ιανουάριο που την ενέκρινε το Κοινοβούλιο σχετικά με τη θερινή ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εναρμονίζεται και το ημερολόγιο για το πότε αλλάζει η ώρα στην Ευρώπη. Ωραία οδηγία είναι. Και είναι η ενάτη οδηγία από τη δεκαετία του 80 που εγκρίθηκε η πρώτη. Και το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια έκθεση ε, αξιολόγησης και με βάση τις πληροφορίες που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε ότι η θερινή ώρα και η χειμερινή δεν έχει αρνητικό ε, αντίκτυπο και οδηγεί σε κάποια εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν θα πρέπει να ανησυχούν τα κράτη-μέλη καθόλου ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα κράτος μέλος δεν έχει ζητήσει από τότε που ε, δημοσιεύθηκε η έκθεση τροποποίηση των σημερινών διευθυντήσεων. Εγώ είμαι ο πλέον αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό, όχι επειδή είμαι αρμόδιος για τις μεταφορές, αλλά ήμουν ε, στην κυβέρνηση της Εστονίας που έκανε ακριβώς αυτό που υπονοείται. Ε, το, πρώτον, ε, το 99 με 2000 καταργήσαμε τη θερινή και τη χειμερινή ώρα. Το αλλάξαμε. Αφήσαμε μία ώρα όλο το χρόνο. Και στη συνέχεια το 2002 επιστρέψαμε στο σύστημα αυτό και επαναφέραμε τη θερινή ώρα. Δηλαδή είμαι ο κατάλληλο άνθρωπος να σα απαντήσω. Έχω προσωπική πείρα. Και ε, δύο δυσάριστα τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αλλαγή αυτής. Και το 2000 ε, το έκαναν αυτό το θέμα πάρα πολύ ε, αντιλαϊκό. αν δεν αλλάξει η ώρα, ε, σκοτεινιάζει πάρα πολύ νωρί και, ε, και ξημερώνει πολύ νωρί. Αλλά το πριν τι να το κάνει το φω τόσο νωρί. Μέχρι να έρθουν τα παιδιά σου από το σχολείο να τα δει, νυχτώνει. Και δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο αυτό στην Εστονία. Και το δεύτερο ήταν ότι υπήρχε πλήρη σύγχυση σε ό,τι αφορά τα ορολόγια, προγράμματα, τα χρονοδιαγράμματα, τα ωράρια και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε για τι μετακινήσει και τα ταξίδια σε άλλε χώρε. Οπότε επαναφέραμε το σύστημα που ισχύει τώρα για τη θερινή ώρα. Εντάξει, δύο φορέ το χρόνο αλλάζουμε το ρολόι. Γυρνάμε το ρολόι και ο κόσμο ευχαριστημένο. Δεν υπήρχε ε, πλέον κανένα πρόβλημα και έληξε αυτό το θέμα, εν πάση Ευχαριστώ πολύ. 7 και 35 η ώρα έχουμε ξεπεράσει. Ναι, ναι, το ξέρω. Ε, την ώρα μα θα σα παρακαλούσα τώρα το εξή. για να επιταχύνουμε λίγο τα πράγματα. Μπορείτε να απαντήσετε γρήγορα σε μια συμπληρωματική που θα σας κάνει ο κύριος Βλόσεβιτς και να ε, απαντήσουμε σε δύο ακόμα ερωτήσεις και τέρμα. Μίτσελ και Χάρκιν, χωρίς όμως πλέον συμπληρωματικές ε, ερωτήσεις. Έχετε το λόγο, κύριε ε, Βλόσοβιτς. Αν θέλετε να κάνετε συμπληρωματική ερώτηση, αν δεν θέλετε μην κάνετε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Επίτροπε. Εγώ έχω μια σαφή αμφιβολία Διότι αν πάρει κανεί το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, βρίσκεται σε διαφορετική χρονική ζώνη από την υπόλοιπη υπηρετική Ευρώπη. Τα ρολόγια δεν είναι στην ίδια ώρα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν τα ρυθμίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Από την άποψη λοιπόν των μεταφορών δεν είναι πολύ καλή ιδέα να ενοποιήσουμε τις ατρακτούς τις ε, ρολογιακές. Επίτροπε, από προσωπική εμπειρία δεν νομίζω ότι το σύστημα πρέπει να το ξαναλλάξουμε. Να αλλάξει το εφιστάμενο σύστημα. Συμφωνώ ότι μπορεί να είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Η επόμενη ερώτηση προς την κυρία Ρέντινγκ. Η πρώτη ερώτηση από τον κύριο Μίτσελ. Παριθμόν 37 για την οσορροπία ελευθερία ασφάλεια. Και η τελευταία θα είναι 38η από την κυρία Χάρκιν. Πράσινη βίβλο για τον εθελοντισμό. Όπω είπα, δεν θα υπάρξουν συμπληρωματικέ ερωτήσει εδώ. You Εντάξει, κυρία Χάρκιν, εσείς ναι, οι υπόλοιποι όχι. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, Βιβιάννη. Hmm. Έχετε το λόγο για την απάντηση. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με περιμένατε για την προστασία και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να εντοπίζουμε καμία αντίφαση ω προ την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Οι αντιτρομοκρατικέ ενέργειε θα πρέπει να διεξαγάγονται σε πλήρη σεβασμό του κράτου του δικαίου και σε πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όπω αυτά καθορίζονται στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με εξισορρόπηση ή με συμβιβασμό των μεν και των δε, πρέπει και τα δύο να τα επιδιώξουμε ως στόχους. Η συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν παρεμποδίζει την ε, έγκριση αποτελεσματικών μέτρων ασφαλείας. Αυτό το αναφέρει και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εγγυηθούν ότι θα χρησιμοποιούνται όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της θερμοκρατίας σε πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα ισορροπίας και όχι εξισορρόπησης των μέτρων ασφαλείας και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κύριε Μίτσελ, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο. Αλλά εξ όσων καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι το ίδιο να αντιμετωπίζουμε του τρομοκράτε και του εγκληματίε, ούτε αυτό με ανησυχεί. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι εμεί ω βουλευτέ δεν δίνουμε αρκετή έμφαση ούτε στη επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε των κρατών μελών το τι περιμένουμε να γίνει ώστε να προστατεύουμε το κοινό να ξέρει κάθε πολίτης ότι προστατεύεται, ότι ο δυτικό του βίο γίνεται σεβαστός, ότι δεν μπορεί ανα πάσα στιγμή να παρισπίσει στο δυτικό του βίο το κράτος. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, είναι σημαντικό κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστούμε η Επίτροπο. Δεν θα μπορούσα παρά να υπερθεματίσω όσα λέτε. Ξέρετε και από την ακρόασή μου πριν λίγο καιρό και από τη δράση μου ως Επιτρόπου των Τηλεπικοινωνιών για την προστασία των δεδομένων, το θέμα αυτό είναι από τα πρώτα σημεία στις προτεραιότητές μου. Κατάφερα να έχουμε αναθεώρηση της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων του 1995 και προκειμένου να προσαρμοστούμε στις εξελίξεις της τεχνολογίας στον κόσμο μας, αλλά επίσης κατέστησα σαφές ότι Άλλο είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία και άλλο τα ιδιωτικά δεδομένα των πολιτών και των προσώπων να μοιράζονται από εδώ και από εκεί. Δεν μπορούν να πληγούν τα προσωπικά δεδομένα και τα θεμελιώδη δικαιώματα λόγω άλλων μέτρων. Καταλαβαίνω γιατί επιχειρηματολογήσατε για το θέμα αυτό και γιατί, για το SWIFT και γιατί ψηφίσατε για το θέμα αυτό. Εμεί τι απόψει του Κοινοβουλίου θα τι λάβουμε σοβαρά υπόψη στην Επιτροπή, ετοιμάζοντα τη νέα μα εντολή για να έχουμε μία νέα συμφωνία SWIFT με, σε συνεργασία με του Αμερικανού μα εταίρου, μια συμφωνία που θα προστατεύει τον ιδιωτικό βίο και θα συμβάζει την ανάγκη αυτή με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Επόμενη και τελευταία ερώτηση, η ερώτηση 38 από την κυρία Χάρκινη για τον εθελοντισμό. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν την έχω αυτή την ερώτηση. Ωραία λοιπόν, αν δεν έχετε την ερωτήση. Έχω πολλές ερωτήσεις εδώ, αλλά δεν έχω αυτήν. Έχω την 88, την 95 και την 100, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε την 38 δηλαδή. Θα πρέπει να απαντήσετε γραπτός. Ζητώ συγγνώμη κυρία Χάρκιν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε μια δήλωση 30 δευτερολέπτων ε, περιμένω την απάντηση της Επιτρόπου γραπτός. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, έχετε μήπως την απάντηση για την 39? has... Ζητώ συγγνώμη, κάτι πήγε στραβά στην οργάνωσή μας, κύριε Πρόεδρε. Τελώ υποσύγχυση. Έχω κάποιες άλλες ερωτήσεις και όχι αυτές που μου ζητάτε. νομίζω χρησιμοποιούμε διαφορετική αρρύθμιση. Η ερώτηση από την κυρία Χάρκιν ήταν για την πράσινη βίβλο για τον εθελοντισμό. Και του κυρίου Πόσελτ. Έχω την ερώτηση του κυρίου Πόσελτ. Κυρία Χάρκιν, να κάνετε μια σύντομη δήλωση και μετά θα ακούσουμε την ερώτηση του κυρίου Πόσελτ και θα ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Ελπίζω ο Επίτροπος να εξετάσει αυτό που πρότεινα, τη δυνατότητα ε, το 2011 που θα είναι Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού να εξετάσουμε και τη δυνατότητα να έχουμε μια πράσινη βίβλο μετά από διαβούλευση με τις ομάδες που ασχολούνται με τον εθελοντισμό και να λάβουμε υπόψη και τη σημασία του να χρησιμοποιήσουμε είτε το εγχειρίδιο του ΟΗΕ είτε το σχέδιο μέτρησης ε, του ΙΣΔΟΕ. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε γιατί δεν έχετε την ερώτηση, αλλά ε, θα λάβετε γραπτή απάντηση. Ευχαριστώ για τη δήλωσή σα Να περάσουμε τώρα στην τελευταία ερώτηση του κυρίου Πόσελτ για τις μειονότητε που είναι κατά εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έχετε. Ναι κύριε Πρόεδρε και μπορώ να διαβεβαιώσω και την ε, κυρία Χάρκιν ότι το θέμα του εθελοντισμού που είναι πολύ σημαντικό ε, απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λάβετε και τις απαντήσεις σε αυτό που μας έχετε ζητήσει. Όσον αφορά τώρα τις μειονότητες που είναι κατά παράδοση εγκατεστημένες, γνωρίζετε ότι αυτή είναι μία από τις αξίες στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σεβασμός δηλαδή ε, των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας αυτό αναφέρεται ρητός στο άρθρο 2 της συνθήκης. Το άρθρο 21 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απαγορεύει ρητός οποιαδήποτε διάκριση ε, για λόγους γλώσσας ή ε, υπηκότητας εθνικής μειονότητας. Ακριβώς λοιπόν ε, αυτό είναι που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάρκεια της θητείας της να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα ακόμα και όταν εφαρμόζεται από κάποιο κράτος μέλος το ευρωπαϊκό δίκαιο. Υπάρχουν μια σειρά από προγράμματα τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες αυτής της μορφής και θέλουμε να συνδυάσουμε τα διάφορα μέσα για να μειώσουμε τις δυσκολίες και τις διακρίσεις που μπορεί να πλήξουν άτομα τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένε μειονότητε. Γνωρίζετε επίσης ότι υπάρχει και νομοθεσία κατά των διακρίσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ίση μεταχείριση ε, ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε και μια πρόταση για μια νέα οδηγία η οποία είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή που θα αυξήσει την προστασία κατά των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ε, πεπιθήσεων, αναπηρίας, ε, σεξουαλικού προσανατολισμού και αφορά και σε άλλα θέματα εκτός της, ε, του χώρου εργασίας και της απασχόλησης. Επίσης υπάρχουν ε, προγράμματα για την καταπολέμηση συγκεκριμένων ε, μορφών βίας και ξενοφοβίας και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι και η λεκτική βία και τα αδικήματα μίσους θα τιμωρούνται σε όλα τα κρατη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή αυτής της απόφασης πλαίσιο όσο το δυνατόν στενότερα και έχει δημιουργηθεί και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ακριβώς για αυτό το σκοπό. Υπάρχει επίσης η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που ε, βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκπλήρωση των καθηκόντων της και υπάρχει και ε, η Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και την Προστασία των Μειονοτικών Γλωσσών. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι ελπίζω ε, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτών που έχουν ήδη υπογράψει και κυρώσει αυτές τις πολύ σημαντικές συμβάσεις. Κύριε Πόσελ, 30 δευτερόλεπτα. Κύριε Επίτροπε, αυτό το τελευταίο ε, αφορά ακριβώς αυτό που με ενδιαφέρει εμένα έχετε έργα για θετική διάκριση και, και μέσα. Θετική διάκριση υπέρ των μειονοτήτων που είναι εγκατεστημένες ε, εδώ και πολύ καιρό κατά παράδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι αρμόδιος και ο οργανισμός των ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων στη Βιέννη. Και πώς οργανώνεται η επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Οι παραδοσιακές μειονότητες παίζουν ρόλο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ε, ε, άδικο από την ίση μεταχείριση ανίσων καταστάσεων. Ε, ευχαριστώ με τον αξιότιμο κύριο Βουλευτή ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο από την ίση μεταχείριση ανίσων ομάδων καταστάσεων. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα σπάνια κονδύλια που διαθέτουμε και τα περιορισμένα με τρόπο πολύ ενεργό και ευφύ. Ε, ε, ο Οργανισμός Εμελιδών Δικαιωμάτων έχει κάποιους στόχους βεβαίως να εκπληρώνει. Αλλά εάν το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσουν από τον οργανισμό αυτό να ε, ανταποκριθεί και σε άλλα καθήκοντα, σίγουρα θα το πράξει. Θα παρακαλούσα τον αξιότιμο βουλευτή λοιπόν να μου διαβιβάσει τα ζητήματα που τον απασχολούν και τις ερωτήσεις που θέλει να θέσει ε, στον ε, Οργανισμό Ανθρωπίνων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα δω τι μπορεί να γίνει ε, για να δώσουμε θετική συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κύριε Ταραμπέλα, μια που ήρθατε, κλείνουμε εδώ τη συζήτηση. Αν θέλετε να κάνετε μια σύντομη τοποθέτηση 32 δεύτερα και με βέβαιος θα απαντήσει και η κυρία ε, Επίτροπος, γραπτός όμως. Αν θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση προφορική εσείς τώρα. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνω ε, τις σχολίες που, ε, ο χρόνος θα χρειάζεται μια ειδική χρονιά αφιερωμένη στη βία κατά των γυναικών που είναι πολύ συχνά ταμπού ακόμα. Πολλές γυναίκες υφίστανται βία και σωματική και ελεκτική και ε, ψυχολογική και συχνά στην οικογένεια και ε, ε, ντρέπονται να το ομολογήσουν. Αν αφιερώσουμε ένα έτος σε αυτή την κατάσταση θα μπορούσαμε να φροντίσουμε αυτό το θέμα να υποχωρήσει από ταμπού και να βγει στο φως και να μπορούμε να αγωνιζόμαστε καλύτερα κατά της βίας κατά των γυναικών. Ευχαριστώ εσάς όλους και την Επίτροπο και τους διερμηνείς. Καλή σας όρεξη.